με το προτινόμενο από την Κομισιόν Προπολογισμό. Όμω, ε, το κείμενο το οποίο διαπραγματεύτηκε ο εισηγητή ε, για τα δύο τάμια ε, είναι κατεμέ το βέλτιστο δυνατό υπό τι παρούσε συνθήκε. Παρακαλώ λοιπόν όλοι να καταψηφίσουμε οποιαδήποτε τροπολογία θα είναι κατά αυτού του κειμένου. Ω εισηγητή, εγώ ήθελα να υπάρχει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παραμένω στην απόψη μου και σήμερα. Αλλά οι στόχοι ε, να εμποδιστούν επενδύσεις σε τομείς όπως είναι η συμπαραγωγή ενέργειας ή η μαζική αστική θέρμανση. Ε, δεν είναι θετικές. Επίσης, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, αλλά αυτά τα λένε ε, κάποια από χώρε που ωφελήθηκαν από τις δραστηριότητες αυτές και τώρα δεν θέλουν να αποφεληθούν άλλα κράτη. Σε αυτή την πρόταση δεν είμαι υπέρ. Ταυτόχρονα προωθούν ε, αγωγούς όπως ο Nord Stream 2 για την παροχή κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Μέρος ε, των Ευρωπαίων Συνταρρυτικών, ο κύριος Φίτο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή και προς όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν στην Επιτροπή για ένα θεμελιώδες κείμενο. Σημερίζομαι την αρνητική σκέψη όλων των συναδέλφων σε σχέση με τις περικοπές που ε, δεν αποτελούν πρόκριμα για μία θετική εξέλιξη. Και θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της ε, της αντίδρασης και δράσης περισσότερο. Δηλαδή τι θα γίνει με τους πόρους μετά το 2021. Αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να ξεπεράσει τις καθυστερήσεις του παρελθόντος σε σχέση με τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις δαπανών, πιστώσεις πληρωμών. Και τέλος το θέμα που σχετίζεται με την ευελιξία για να γίνει καλύτερη χρήση αυτών των πόρων σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ από τους φιλελεύθερους, Κύριε Μιχαήλοβα. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη συμβολή τους στο έργο υπέρ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής. Συνεργαστήκαμε με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και ιδίω συνταχθήκαμε υπέρ ε, περισσότερης ευελιξίας, αποτελεσματικότητας, απλούστευσης των ε, διαδικασιών των δύο ταμείων. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό να συνεχίσει να στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα θετικά. Πρώτα απ' όλα, η αυξανόμενη συμβολή των ταμείων στην επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, μείωση 40% των εκπομπών. Επίσης, πολλές προτάσεις της Επιτροπής Ρέτζη πέρασαν με αντικείμενο την ενίσχυση της αστικής διάστασης του θέματος. Για να υλοποιήσουμε δηλαδή και το θεματολόγιο για τις πόλεις. Είχαμε όμως και άλλα θετικά στοιχεία μεταρρύθμισης, την αλληλεπίδραση με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε κατά τα άλλα την θεματική στόχευση, την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα των περιφερειών. Σε άλλα σημεία, η έκθεση καλεί επίσης για μια Ευρωπαϊκή Ένωση χαμηλότερων εκπομπών και γι' αυτό αποκλείουμε και κάποιου τομείς, σχετικούς τομείς από τη χρηματοδότηση. Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους με βάση σαφή κριτήρια αποκλεισμού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, από την Σκρέλτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε μάλλον όλοι μας ότι το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ είναι πολύ σημαντικά για τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν οι χώρες να σημειώσουν πρόοδο στις περιφέρειες όπου ε, υπάρχει υστέρηση έτσι και αυτέ οι περιφέρειες θα έρθουν πιο κοντά στις πιο αναπτυγμένε χώρες. Αξιοποιούμε λοιπόν κονδύλια για να επενδύσουμε στις κοινέ μας αξίες. Ως ο όμω όμως είμαι κάπως απογοητευμένο από τα αποτελέσματα εν γέννη. Μπορούσαμε και καλύτερα και τούτο διότι ξόδεψαμε πολλά για επενδύσεις ας πούμε στα ορυκτά καύσιμα, στι υποδομές για το φυσικό αέριο. Πράγματα τα οποία δεν θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτικών που ήδη έχουμε συνομολογήσει. Με τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας δεν θα μπορέσουμε, φοβάμαι, να αξιοποιήσουμε σωστά τα κονδύλια για τους σωστούς σκοπούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα εκ μέρους της Κυρία Μιχέλης. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πράγματι ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι και παραμένει ένα πολύ λογικό εργαλείο υποστήριξη ιδίω τη υπαίθρου και εμείς ε, είμαστε υπέρ ε, της κοινωνικής εξίσωσης όλων των περιφερειών. Πρέπει τώρα να εστιάσουμε σε μια πιο πράσινη Ευρώπη και αυτό γίνεται σε αυτή την έκθεση και είναι θετικό. Όμως δεν θέλουμε μόνο διακοσμητικά μέτρα. Θέλουμε εκ των βάθρων οικολογική κοινωνική αλλαγή. Θέλουμε να είναι σαφές το εξή. Ε, χρειάζεται αλλαγή θεώρησης και διατροτικές διαρρυθμίσεις. Ε, αυτό όμως ε, το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε με 40% ε, των επενδύσεων για την οικολογική κοινωνική μετάβαση, για τη δίκαιη μετάβαση όπως λέγεται. Επίσης δεν είμαστε υπέρ ε, του ότι σε έναν φιλόδοξο κατάλογο αυτών των αλλαγών κοινωνικών οικολογικών θα υποστηρίζουμε επενδύσεις ε, σε αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη που θα φιλοξενούν low cost εταιρείες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουμε σχέδια εντάξει τα οποία δεν θα λαμβάνουν υπόψη ε, την καταγωγή, παράδειγμα, των μεταναστών. Η αλλαγή διαρθρωτική στο κοινωνικό και οικολογικό πεδίο θα πρέπει να συνδιαμορφωθεί με ενεργό τρόπο από τους πολίτες και γι' αυτό ε, υποστηρίζουμε αυτά ως γκουε ως, από το η κυρία Νταμάτ. E Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κλείσει η πρώτη ανάγνωση για τα ταμεία έτπα και συνοχής. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διασπάθηση χρήματος δυνάμει του ε, συμφώνου και επίσης να μην γίνεται χρήση ορυκτών καυσίμων. Πώς μπορούμε να πούμε ότι για πολλωστή φορά αρνηθήκαμε αυτά τα κονδύλια, πώς μπορούμε να ε, δεχτούμε τα λεγόμενα των νέων με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των αλλαγών του κλίματος, εάν δεν έχουμε μία οικονομία ε, επανακατανομής, ιδιαίτερα για τα ορυκτά καύσιμα. Θα ήθελα όλοι να υποστηρίξετε τις τροπολογίες για το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στούχερα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΤΠΑ έχει έχει μεγάλη σημασία και στην ουσία ε, τι κάνουμε. Ε, ε, μεταβιβάζουμε τα χρήματα του φορολογουμένου σε ένα ταμείο που δεν αποφέρει καρπούς. Και δεν σημαίνει αυτό ότι τα χρήματα μεταφέρονται από τους πλούσιους, τους φτωχούς. Απλώς τα, παίρνουμε τα χρήματα από τη μεσαία τάξη και τα μεταφέρουμε στους υπερπλούσιους της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ένα στρατό δικηγόρο και ξέρουν πολύ καλά πώς να διαχειριστούν ε, αυτά τα χρήματα και τον πλούτο. Ο φορολογούμενος είναι το απόλυτο θύμα και αναρωτιέμαι πότε θα σταματήσει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης. Α, μάλλον κύριε Στούχερ, θα δεχτείτε μπλε κάρτα από ένα συνάδελφό σας. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Νίστελ Ρόι έχει το λόγο. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που ο κύριος Στούγκερ μίλησε για σχέση αιμομιξίας ε, μεταξύ ΕΤΠΑ και μεταφοράς ε, αυτό με άφησε εμβρόντιτο, γιατί στη Ρέτζη δεν ήταν ποτέ παρόν όταν συζητήσαμε το θέμα. Και τα, οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται υπέρ των ε, φτωχών. Πώς μπορείτε να λέτε κάτι τέτοιο. Διαβάστε τα έγγραφά σας. Μπορείτε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω κι εγώ ευθέως, όσο ευθέως με ρωτήσετε. Εσείς στη Ρέτζη, στην ουσία στέλνετε τα χρήματα των ε, φτωχών στους πλούσιους. Ε, δηλαδή, ε, εγώ βρισκόμουν τότε στη Ρουμανία. Μιλήσατε για δημιουργία για, μιλάτε για ανούσιες δαπάνες και θα έπρεπε να ντρέπεστε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης από τους μη εγγεγραμμένους. Τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού για το έτπα και τα ταμεία συνοχής περί καταπολέμησης της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανεργίας. Αυτά κρίθηκαν στην Ελλάδα, όπου τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η Ελλάδα πρότευσε σε απορροφητικότητα των ευρωκονδυλίων και η φτώχεια απογειώθηκε, η μερική ευέλικτη απασχόληση εκτινάχθηκε, βυθίζοντας ακόμα πιο βαθιά στα διέξοδα το λαό γιατί τα ευρωνοσιακά κονδύλια όλα ιδρώτα του λαού από την άγρια φορολαιλασία του κατευθύνονται στην ενίσχυση των ευρωνοσιακών μονοπωλίων. την ίδια ώρα αντιπλημμυρικά αντιπυρικά αντισυσμικά έργα ζωτικές ανάγκες για υγεία παιδεία μένουν ανικανοποίητες με κριτήριο τα κέρδη για τα μονοπόλια και επιπρόσθετα τα πρόστιμα η αιρεσιμότητα ο λογαριασμός μετακυλείεται μέσω χαρατσιών και φορολογίας και πάλι στο λαό. με ισχυρό κκε θα αποκτήσουν πιο δυνατή φωνή οι διεκδικήσει του εργατικού λαϊκού κινήματος στην πάλη για συνολικές ανατροπές έτσι ώστε όλα αυτά τα κονδύλια να χρηματοδοτήσουν έργα κέρια για την ανακούφιση και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ευχαριστούμε πολύ επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Βανίστελ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. Εμείς στην Ολλανδία δίνουμε προτεραιότητα στις πόλεις, δηλαδή να ε, ε, επιδοθούν ένα 10% και όχι 5%. Αλλά πολλοί μίλησαν να 2,4 δις ευρώ για να ενισχύσουμε την ε, κοινοτική συνοχή στις μικρές πόλεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι θα γίνει μια μεγάλη μετακίνηση από τις αγροτικές περιοχές της πόλης. Μιλάμε για 8 εκατομμύρια συνολικά. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι οι ευφυείς ε, κομοπόλεις αυτό το προωθήσαμε και θα το προωθήσουμε και υπό την Φινλανδική και ε, Κροατική Προεδρία. Θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε έπειτα η συγχώνευση των δύο ταμείων θα γίνει το έτπα και το Ταμείο Συνοχής. Η απλούστευση φαίνεται πολύ καλή, αλλά έμπρακτα έχουμε αποδημο... αποδυναμώσει συγγνώμη, αυτά τα ταμεία. Θα πρέπει να μεταφέρουμε γνώση και δεξιότητες, να καινοτομούμε. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ζητήματος και αφορά και την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι θα φτάσουμε σε μια νέα οικονομία 2021-2027. Εγώ σας μιλάω για τελευταία φορά ως Ευρωβουλευτής από την Ολλανδία και ε, ε ισότητα στην Ευρώπη σημαίνει έμπρακτη ισότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μισή που παίρνουμε το λόγο σήμερα το κάνουμε για τελευταία φορά, αλλά να σεβόμαστε όλο τον χρόνο. Κυρία Ροντρίγκη. Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι το Ταμείο Συνοχής δεν βοήθησε τόσο την Ελλάδα όσο και τη χώρα μου, την Πορτογαλία. Άρα με αυτή την έκθεση θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική συνοχής να μειώνει τις ανισότητες και να έχουμε μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και τις περιφέρειες. Υπάρχουν ε, δημογραφικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι εξόχως ε, απομακρυσμένες περιφέρειες δεν ευνοούνται Γι' αυτό το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτές τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό αφορά και τις υποδομές στο αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη θεματική που ισχύει και σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τόμασιτς. η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτούμε απευθείας έργα χωρίς ε, γραφειοκρατικά εμπόδια. Πολλές χώρες, όπως η Κροατία από την οποία προέρχομαι, δέχτηκαν πολύ μεγάλη βοήθεια από το Ταμείο Συνοχής. Ήρθαμε πιο κοντά στις πλουσιότερες χώρες και έτσι οι θέσει εργασία διατηρούνται για ένα καλύτερο μέλλον. Ως μέλο της Επιτροπής Ρέτζε Περιφερειακών Υποθέσεων και Κροάτισα υποστηρίζω τη νέα προσέγγιση, τη μεταρρύθμιση με καλύτερους στόχους, σαφέστερου στόχους που κοιτάζουν το μέλλον για πιο πράσινε και αηφορικέ λύσει. Τονίσω για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να καταργούμε τα περιτά γραφειοκρατικά εμπόδια σε όλα τα επίπεδα. Να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους τοπικούς παράγοντε να βελτιώνουμε τη δημόσια διοίκηση και να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε ακόμη περισσότερο αυτούς οι οποίοι υλοποιούν τα έργα εν τέλει. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και τώρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για πολλές περιφέρειες το ΕΤΠΑ είναι μια νησίδα ελπίδες σε έναν ωκεανό όμως λιτότητες. Γι' αυτό το λόγο το Ταμείο είναι ζωτική σημασία και τις επενδύσει του πρέπει να τι ενισχύσουμε στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες κατά κύριο λόγο. Να αντιταχθούμε λοιπόν στις μειώσεις που πετανεύει η Κομισιόν. α αποκραστήσουμε την, τα ποσά της προηγούμενη προγραμματικής περίοδου. Τώρα για τη συγχρηματοδότηση. Η Κομισιόν σε ορισμένε περιπτώσει ε, προτείνει μειώσει 70%. Εμεί πιστεύουμε ότι η συγχρηματοδότηση πρέπει να ανέλθει στο 85%. Εν ώψη λοιπόν τη νέα περίοδου, δεν είναι δυνατόν να μην συμφωνήσει η Κομισιόν με το Κοινοβούλιο, δηλαδή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τι ε, πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Ευχαριστώ. Και τώρα, κύριος Μπόκοβιτς. Το ΕΔΠΑ και το Συνοχή είναι τα δύο ταμεία τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό είναι και μία από τι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και παραμένει πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην περιορίσουμε λοιπόν τα διαθέσιμα κονδύλια. Αλλιώ η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να πετύχει του στόχου τη. Συμφωνώ απολύτω με του πράσινου στόχου, με την ενεργειακή απόδοση Επίση, με παίρνει τροπολογία. σύμφωνα με την οποία 5%, 2,4 εκατομμύρια πηγαίνουν προ τα έξυπνα χωριά. Είναι αλήθεια ότι πολλοί εγκαταλείπουν την ύπεθρο. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ΕΤΠΑ θα μπορέσει να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να δημιουργήσουμε λοιπόν θέσει εργασία στι περιοχέ, αυτέ, στις αγροτικέ περιοχέ. Και αυτό θα μα επιτρέψει επίσης να έχουμε μια πιο σύγχρονη γεωργία. Αυτός ο τύπος επασχόλησης, αποκεντρωμένο αν θέλετε, και με κοινωνικό χαρακτήρα, μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Το χρωστάμε αυτό στις αγροτικέ περιοχές. Επίση, η αποκεντρωμένη ενέργεια. Όλα αυτά είναι μέτρα υπέρ των έξυπνων χωριών. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η αποκέντρωση είναι ο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζουφρίντα. E ΕΤΠΑ και Ταμείο συνοχή είναι τα καλύτερα μέσα υποστήριξη υποδομών και περιφερειών. Αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε για τις περιφέρειες και αναφέρομαι και στην δική μου Σικελία. Αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά προσκόμματα και δεν ε, μειώνεται πάντα η γραφειοκρατία. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να απογειωθούν συγκεκριμένα προγράμματα γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς η περιφερειακή διάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους αυτούς για να λάβουμε υπόψη και την εδαφική και περιφερειακή διάσταση που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα νησιωτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες υπέρ των πολιτών Μόνο έτσι θα συμφιλειώσουμε τους πολίτες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής τάσσονται υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης για την μείωση των χασμάτων μεταξύ περιφερειών. Όμως θα πρέπει να είμαστε σωστοί και να δεχτούμε τα ε, ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε υπέρ αυτών των δικτύων ευρυζωνικής ε, μεγάλης ε, υψηλής ταχύτητας και να προσελκύσουμε και τους ιδιωτικούς επενδυτές και να έχουμε και μεταφορά αποτελεσμάτων in situ. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία μεταξύ εταίρων στα πλαίσια αυτής της διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λουί Ζωζεφ Μανσκούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ Συμφωνώ με όσους συναδέλφους επένεσαν το έργο του εισηγητού. Το κείμενο της Επιτροπής ΡΕΚΙ νομίζω ότι είναι σωστό μεταξύ άλλων συμβάλλει στην επαναπεριφεροποίηση ε, και ελαστικοποίηση των ταμείων ε, συνοχής περιφερειακής ανάπτυξης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και για καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. Επίσης, ε, πολύ θετικέ είναι οι προτάσεις που διατηρούν τη θεματική συγκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί έτσι ελπίζω ότι θα προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή και θα είναι κοντά στην κάλυψη των αναγκών των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Ιδίως επειδή προέρχομαι από μια γαλλική εξόχως απόκεντρη περιοχή, χαίρομαι που υπάρχουν πιο εξειδικευμένα μέτρα ε, που ε, θα χρηματοδοτήσουν ε, τις ε, υποδομές σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες για τις οποίες το ΕΤΠΑ είναι πολύ σημαντικό. Κλιματική περιβαλλοντική στόχη είναι προτεραιότητα, γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα μας προς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μοντέρο Δεαγιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ουσία το ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής είναι ταμεία ζωτικής σημασίας για τις περιφέρειες, αλλά ιδιαίτερα για τις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες. Η κυρία Κορίνα Κρέτσου, η Επίτροπος, δεν μας μίλησε για τις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε αναφέρεται σε αυτές. Θα θέλαμε να μην δεχτούμε περικοπές στην πολιτική συνοχής παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν λαμβάνουμε υπόψη περιφέρειες όπως αυτή της Μαδέρας και δεν προωθείται καινοτομία, απασχόληση, στέγη, ένταξη μεταναστών και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια συμφωνία αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να δεσμευτούν και τα κράτη σε σχέση με τα τελικά ποσά για να έχουμε μια καλύτερη πλαισίωση των εξόχως απομαξμένων περιοχών. Ο κύριος Πίτσουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Ταμείο Συνοχής είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πρόθεση της ε, εδαφικής κοινωνική ε, συνοχή μεταξύ των περιφερειών και είναι και μεγάλο επίτευγμα της Ένωσης η νέα πρόταση. Περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία για να προσαρμοστούμε στο μέλλον. Υπάρχουν λοιπόν μέτρα που θα καταστήσουν απλούστερη τη χρήση των κονδύλων των ταμείων. η αύξηση ε, του βάρους ε, συγχρηματοδότησης ε, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολο το να υποβάλουν υποψηφιότητα για έργα. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Θέλουμε περισσότερη ευελιξία, μεγαλύτερες δυνατότητες για τις δημόσιες διδικήση ε, μέλλον ε, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχή, θα ε, εξασφαλιστεί μόνο με επαρκή προπολογισμό. Λόγω του Brexit και τη απροθυμίας κάποιων κρατών μελών να βάλουν λεφτά, τα πράγματα δυσκολεύουν για αυτά τα δύο ταμεία. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το 174 που θα περιλάβει και τα νησιωτικέ περιοχές. Η κυρία Βέστφαλη τώρα το λόγο. Κέρστιν Βέστφαλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θεωρώ ότι είναι κρίμα ε, που έφυγε ο μια εγγεγραμμένο συνάδελφο, γιατί έπρεπε να άκουγε ε, τι ε, λέμε και να μην λέει τόσε ανοησίε όσε είπε. διότι το πρόγραμμα εξασφαλίζει την ανάπτυξη για όλου, για όλε τι ε, περιφέρειε, για όλου του πολίτε. Θέλουμε να επενδύσουμε σε μια σύγχρονη ψηφιακή, πράσινη, κοινωνική Ευρώπη. Την Ευρώπη ε, των ανθρώπων. Είτε ζουν στην πόλη, είτε ζουν στην Ήπεθρο. Θέλουμε να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία, τι νέε θέσει εργασία, την καταπλέμψη τη κλιματική αλλαγή. Και πρώτων ευρωεκλογών είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, το Ταμείο Συνοχή, το ΕΤΠΑ, είναι το 1 τέταρτο του προπολογισμού. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό στον κόσμο. Τα χρήματά του γυρίζουν πίσω, γυρίζουν στι περιφέρειε, γυρίζουν στι πόλει του. μάλιστα ε, είναι δαπάνε πολύ λογικές. Δεν θέλουμε να ε, τονίσουμε, δεν θέλουμε να στηρίξουμε μάλλον και να επενδύσουμε σε αεροδρόμια φαντάσματα που δεν θα πετάει καμιά εταιρεία. Εμεί θέλουμε ένα ταμείο που θα ε, δοθούν ε, τα κονδύλια εκεί που χρειάζεται για να είναι σε καλή κατάσταση η Ευρώπη για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρθία Πέρεθ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε εγκρίνει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα είχα την τιμή να είμαι εγώ η, εισηγήτρια για το πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση των δημογραφικών προκλήσεων και την καταπολέμηση της απερίμωσης. Σήμερα, με την έγκριση του κανονισμού για το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δίνουμε σάρκα και οστά σε κάποια εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την απερίμωση. Και χάρη στι τροπολογίε, στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι τουλάχιστον 5% του Ταμείου θα πρέπει να δίνεται σε ζώνες με δημογραφικά μειονεκτήματα. Και το άρθρο 10 περιλαμβάνει την δυνατότητα ειδικών κονδυλίων στις συμφωνίες σύνδεσης, ε, σύνδεσης για να καταπολεμήσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό για την υπεθρό μας ε, η ευρωπαϊκή πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής να δίνουν ελπίδα στους λαούς που δυνοπαθούν αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, χαιρετίζουμε το νέο κανονισμό που δείχνει ότι είναι ευαίσθητος απέναντι στις δημογραφικές μας προκλήσεις. ευχαριστώ. Περνούμε στο Catch τώρα. Μια και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα σας πρότεινα να ακούσουμε τρεις από κάθε ομάδα που ζήτησε το λόγο στο Catch the Eye, για μεγαλύτερες. Ο κύριος ε, Μιγενμόν, το ΦΕΝΤΕΡ είναι πολύ σημαντικό όργανο και εργαλείο για να δοθεί έμφαση στη συνοχή στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και θα ήθελα να σταθώ σε ένα πρόβλημα που πλήττει τη Γαλλική, τη δική μου γενέτειρα. Κυρίω ε, αναφέρομαι στη γύρωση του πληθυσμού και στη φθήνουσα πορεία που έχει πάρει η δημογραφική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση τη ε, Γαλλικία έχει ε, λάβει κάποια θετικά μέτρα και μάλιστα προωθεί και ένα σχετικό νομοσχέδιο για τη δημογραφική ανάπτυξη. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντείνουν τι προσπάθειέ του. Και η δημογραφική μείωση θα πρέπει να είναι σημαντικό κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων και με τον κύριο Βαλκάθελ Σίσο κατέθεσαμε πολλές τροπολογίες και συγκεκριμένα άρθρα και κυρίως το 10α που μιλάει για ζώνες με δημογραφικές προκλήσεις ώστε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε δήμους και κοινότητες που υποφέρουν από την απερίμωση. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα εδάφη να υφίστανται σε ειδικά σχέδια για να τονίζεται χάρη στην αύξηση των επενδύσεων η δημογραφική ανάπτυξη. Και μάλιστα και στι συμφωνίε σύνδεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπει ειδικά κονδύλια για να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικέ προκλήσει στι χώρε τη σύνδεση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μιγιανμόν. Ο κύριο Χωσέ Μπλάνκο Λόπε έχει το λόγο τώρα. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε αν υπάρχει μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αξία της ελληνικής η αξία αυτή, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παλιδρομήσει επουδενή στις πολιτικές που δίνουν περιεχόμενο, άρκα και οστά στην απαραίτητη σύγκληση μεταξύ των περιφερειών. Χαιρετίζω τι βελτιώσει που επιφέραμε στον κανονισμό με τι τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δημογραφικό ζήτημα. Θα πρέπει να αφιερώσουμε κονδύλια για να καταπολεμήσουμε την απερίμωση, να καταπολεμήσουμε τη γύραση του πληθυσμού που πλήττει την οικονομική αναζωογόνηση και την επιβίωση του ε, της Υπήρου μας. Από αυτό εξαρτάται η επιβίωση του κοινωνικού μας μοντέλου και της κοινωνικής και δαφικής συνοχής. Χαίρομαι που δίνουμε περιεχόμενο στην ε, συνεκτική και κοινωνική Ευρώπη που προσπίζουμε οι περισσότεροι. Είμαστε υπέρ τη ισότητα, τη ε, εδαφική και κοινωνική συνοχή. Αυτό ήταν ανέκαθεν το λάβαρό μα και εμβληματική μα προσπάθεια. Ιδιαίτερα για περιοχέ όπω τη, τη, τη γενέτειρά μου, τη Γαλλική. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η σχετική συμφωνία. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστοφ Χέτμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αναφυσβήτητο ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής είναι τα, από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιήσουμε μια ουσιαστική οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξίσωση των ανισοτήτων, ε, η απάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό, χάρη στα, στα κονδύλια αυτά, στηρίζουμε την ε, ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και στα αστικά κέντρα και, στις, και στην Ήπεθρο. Ε, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτό το έγγραφο που τονίζει την ανάγκη σημαντικών επενδύσεων. Χρειάζεται επίση μεγαλύτερη ελαστική, ελαστικότητα στην επιλογή των κριτηρίων επενδύσεων. Χάρη σε αυτό, τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειε θα μπορούν να αποφασίζουν ποιε είναι οι επενδύσει που ανταποκρίνονται καλύτερα στι ιδιαίτερε ανάγκε του. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Χέτμαν. κυρία Κέρτον Τάρλινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το Σάββατο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έκαναν πορεία και ζήτησαν ε, νέο δημοψήφισμα για τον Brexit. Μεταξύ αυτών και πολλοί άνθρωποι από τη δικιά μου περιφέρεια, την βορειοανατολική Αγγλία, καθώς ε, φαίνεται πως η πραγματικότητα του Brexit πλέον γίνεται αντιληπτή, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Η περιοχή μου έχει ωφεληθεί από τις μεγάλες επενδύσεις από το ΕΤΠΕ. Ένα δισεκατομμύριο λίρες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το 2014-2020. Ζωτικοί πόροι που δημιουργούν δουλειές, αναβαθμίζουν τις υποδομές και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά είναι λεφτά των Βρετανών φορολογουμένων ούτως ή άλλως. Ναι, είναι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέμει με βάση την οικονομική ανάγκη και όχι την πολιτική προτίμηση. Είναι η αλληλεγγύη στην πράξη. Αν παραμείνουμε, η Βορειοανατολική Αγγλία έχει εγγυημένα εκατομμύρια λίρες. Αν βγούμε, είμαστε στο έλεος του Westminster. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει κάποιους όρους περί Brexit. Σας παρακαλώ να μην τους χρησιμοποιήσουμε και να μείνει η Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ιβάνα Μάλετιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι μίλησαν για τα πλεονεκτήματα του ΦΕΝΤΕΡ και του Ταμείου Συνοχής και πόσο βελτιώνουν αυτά για τη θημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Με τη νέα πρόταση έχουμε μια πολύ σημαντική διάταξη γιατί επιτρέπει την, τις σημαντικές υποδομές στα κράτη-μέλη και την αύξηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένες περιφερειακές επενδύσεις ε, για την περιφερειακή ανάπτυξη και επίση ε, κάποιες ελάχιστες επενδύσεις για την αγροτική ανάπτυξη. Είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύση, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν μιλούμε για τα ευφύ χωριά, αν μιλούμε για αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, αν μιλούμε για την σημασία που έχει η ισορροπημένη ανάπτυξη στην Ευρώπη για εξίσου του βιωτικού επίπεδου και ανήψη του βιωτικού επίπεδου όλων των κατοίκων, θα πρέπει να προβλέψουμε χρηματοδοτικά μέσα από τον κοινοτικό προπολογισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο νέο κανονισμό, ανταποκρίνεται στι ανάγκε των συμπολιτών μα και θα συμβάλλει σε εξισορροπημένη ανάπτυξη των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριο Χουάν Λόπε Αγγιλάρη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε Γιώροβα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το καθήκον του, δείχνοντα πυγμή και αναλαμβάνοντα τι ευθύνε του για πολύ σημαντικού κανονισμού για το Ταμείο Ανάπτυξη, ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και ε, το Ταμείο Συνοχή, ε, αφιερώνοντα ένα τέταρτο του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ για, το για την περίοδο 2021-2027. Έχουν σημαντικά αυτά τα μεγάλα κονδύλια, κυρίω για τι μειονεκτού περιοχέ και έχει κέρια σημασία για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ, για τη διασυνδεσιμότητα, για τι μεταφορέ, για τη συμπερίληψη στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Τώρα, μία εγγύηση για την ε, καταπολέμηση των προκλήσεων των κλιματικών αλλαγών. Να λαμβάνεται υπόψη ε, και η προστασία του περιβάλλοντος και η κυκλική οικονομία όταν μιλούμε για τη διαχείριση των αποβλήτων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε καμία εξαίρεση από τη συμβαστική λύση, ότι δεν χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά κανένας αποτεφρωτής για τη διαχείριση αποβλήτων, αν δεν υπόκειται στην αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που ε, δήλωσαν συμμετοχή, αλλά ακριβώ επειδή στις 12.30 αρχίσουμε ψηφοφορίες δεν ε, έχουμε χρόνο για ένα ακόμη θέμα. Ε, και γι' αυτό δεν μπόρεσα να δώσω το λόγο σε όλου που ζήτησαν τον λόγο για το Κατστιάι. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σήμερα μιλήσαμε για κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για τον επόμενο κοινοτικό προπολογισμό, για την πολιτική συνοχή, για το επόμενο Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ταμείο Συνοχή. Αλλά ταυτόχρονα δεν μιλούμε μόνο για χρήματα. Μιλούμε για πολιτικέ που εδράζονται στην αλληλεγγύη και για πολιτικέ που θα βοηθήσουν τι περιφέρειες ε, και κυρίως αυτές που υστερούν σε σχέση με το ΑΕΠ τους και την ανάπτυξή τους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν αφορά μόνο τα χρήματα, το οικονομικό σκέλος, ο κανονισμός, αλλά δεν είναι αμεληταίο και αυτό το οικονομικό σκέλος. Την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα έχουμε περισσότερα κονδύλια για την πολιτική συνοχή. Και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια κατάσταση θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, ξοδέψουμε σωστά αυτά τα κονδύλια ώστε να πιάσουν τόπο. Και αυτό συζητήσαμε σήμερα. Όλοι έχουμε επίγνωση ότι με λιγότερα κονδύλια έχουμε περισσότερε προκλήσει και θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για να πιάνουν, επαναλαμβάνω, τόπο τα χρήματα, ιδιαίτερα όταν είναι λιγότερα. Θα πρέπει να γίνεται σωστή εκταμείευση των κονδυλίων, ώστε να καταλήξουμε σε έξυπνες και βιώσιμες επενδύσεις. Και φυσικά στο επίκεντρο θα πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος γιατί ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση ε, χάρη σε παιδί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα πρέπει να έχουμε ε, πιο υγιή ποτάμια, καλύτερο περιβάλλον και γι' αυτό οι επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και αυτά τα κριτήρια. Με γνώμονα φυσικά το να πιάνουν τόπο τα κονδύλια ώστε να ωφελούν οι επενδύσει στους Ευρωπαίους πολίτε. Γι' αυτό και έχουμε τη θεματική συγκέντρωση και την ανάγκη για ξεκάθαρη προστιθέμενη αξία των επενδύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, την θετική του συνεισφορά και ευελπιστώ ότι αύριο θα εγκριθεί η θέση της πρώτης ανάγνωσης για το σύνολο του νομοθετικού πακέτου της πολιτικής συνοχής για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την νομοθετική διαδικασία τον Οκτώβριο το αργότερο. Γιατί αν θέλουμε να καθυστερήσουμε τα προγράμματα του 2020, όχι μόνο θα πρέπει να εγκρίνουμε φέτο του αντίστοιχου ε, κανονισμού, αλλά και θα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες έγκαιρα και πρόθεσμα να ετοιμάσουν τα σχετικά έγγραφα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε προτάσει που θα διακυβεύσουν την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των σχεδίων τη πολιτική συνοχή. Και τέλο θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των εφιέστερων ε, πόλεων και χωριών. Ε, αυτό προσπαθεί με, μεταξύ άλλων η πολιτική συνοχή να εξορροπεί την ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών περιοχών και αστικών περιοχών. Και αυτό θα είναι ζητούμενο και στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Και ο κανονισμό περί κοινών διατάξεων περιλαμβάνει ένα νέο στόχο πολιτικής, ε, προωθώντας την βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παράκτιων, υπαίθριων και αστικών περιοχών με τοπικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη πολυτομιακή προσέγγιση για την αστική ανάπτυξη. Με τις στρατηγικές αυτές θα ενισχύσουμε την συνοχή των επεμβάσεων και το στρατηγικό προγραμματισμό και σίγουρα η ανάπτυξη η ανάμειξη των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών θα βελτιώσει την ε, ανάληψη ευθύνη σε αυτό το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ο εισηγητή τώρα, ο κύριος Κοτσολίνο. Νομίζω ότι αύριο πραγματικά θα καταφέρουμε να περάσουμε την έκθεση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία Βλέπετε εδώ πέρα και ακούσατε ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία τη συζήτηση αυτή, φαίνονται άλλωστε και οι στροπολογίε που έχουμε καταθέσει. Όσον αφορά εμένα, θα ήθελα να πω το ακόλουθο, συνοψίζοντα τη συζήτηση αυτή, όσον αφορά το ζήτημα τη θεματική συγκέντρωση. Εμεί ευθυγραμμιζόμαστε εδώ πέρα με τι βασικέ ενδείξει που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό που κάναμε είναι ότι δικαιολογημένα ενισχύσαμε την περιφερειακή διάσταση ακριβώς για να υπάρχει απαραίτητη εξισορρόπηση ως προς την εδαφική συνοχή. Το είπαν αυτό και πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν και στο ε, περιβαλλοντικό, στην περιβαλλοντική διάσταση. Ουδέποτε υπήρχε τέτοια συγκέντρωση σε στόχους περιβαλλοντικού σε τοπικό, περιφερειακό και δαφικό επίπεδο. Έχουμε ξεπεράσει το 30% πλέον των πόρων για τα προγράμματα υπέρ του περιβάλλοντος. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η αρχή που έχουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ευελιξία, την οποία βλέπουμε και στον ίδιο τον κανονισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε καλύτερη συγχρηματοδότηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους δημόσιου πόρους και μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ίδια την πολιτική συνοχή. Εν κατακλείδη νομίζω ότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι έχουμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε καθόλου την ε, πραγματικότητα την οποία βιώνουν πάρα πολλές περιφέρειες τα τελευταία χρόνια, όπου είχαμε δημογραφικές ε, τροποποίησεις, αλλά που είχαμε και μία μείωση, αν θέλετε, της παρουσίας του ίδιου του κράτους, αλλά και της Ευρώπης. Λιγότερες υπηρεσίες, λιγότερες δημοσιονομικές ευκαιρίες. Εκεί ακριβώς θέλουμε να επέμβουμε με το Ταμείο Συνοχής, με την πολιτική συνοχής, για να φέρουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, αν θέλετε, της πρωτοβουλίας αυτής και ελπίζω αυτό θα επιβεβαιωθεί και στην αυριανή ψηφοφορία και ότι η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί και με την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη μας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε και τους, συζητητέ τους εισηγητές για το θέμα αυτό. Τον εισηγητή μάλλον είναι εμφανής η στην προσπάθειά του. Ολοκληρώνεται αυτό το, θέμα και περάμε στο επόμενο την κοινή συζήτηση με θέμα την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και τις διαδικτυακές πωλήσει αγαθών. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Εύελιν Γκέπχαρτ και του κυρίου Άξελ Βος για τη συμβάση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του κυρίου Πασκάλα Ριμόν με θέμα τις συμβάσεις για την πώληση προϊόντων. Πρώτα θα λάβει το λόγο η εισηγήτρια της πρώτης έκθεσης, η κυρία Εύελιν Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε. Σε αυτό το κοινοβούλιο ζούμε πάντα συνεχώς εκπληκτικές στιγμές και στην περίπτωση αυτή είναι ακόμη πιο εκπληκτική αν αναλογιστείτε τη συνεργασία μου με τον κύριο Άξελ Φως το νομοθέτημα αυτό είναι μάθημα για το ότι τα καλύτερα επιχειρήματα προκύπτουν όταν και η αντίθετη πλευρά αναπτύσσει τα δικά της. δύο αυτές δίδυμες οδηγίες κάναν πάρα πολλά για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών χρησιμοποιείται όχι μόνο όταν πληρώνουν οι καταναλωτές με νόμισμα, αλλά και όταν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα για να δείξουν παραδείγματος χάρη στοχευμένες και εξατομικευμένες ε, διαφημίσεις. Βεβαίω, πρέπει να ισχύει άρα και η ίδια προστασία. Είτε κατεβάζουν μια εφαρμογή οι καταναλωτέ ε, και ανεξαρτήτως του εάν ε, γίνονται αυτά μέσω ενό έξυπνου ψυγείου, παραδείγματο χάρη. Όλο το software θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό με το οποιοδήποτε υλικό. Οι καταναλωτές ε, έχουν ε, απέτηση πλέον για αναβαθμίσεις του λογισμικού οι οποίες θα οδηγούν σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ε, των προϊόντων τους ε, χωρίς την οποία βεβαίως καθίστανται άχστα. Η φορητότητα του περιεχομένου επίσης είναι ένα άλλο θέμα το οποίο οι καταναλωτές και καταναλώτριες βεβαίως χρησιμοποιούν σε διάφορες ε, υπηρεσίες ε, και εφαρμογές. Η διατήρηση της ελάχιστης ε, εναρμόνισης με την ταυτόχρονη παράτηση των προθεσμιών καθώς επίσης και η αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως αλλά και η παράταση από έξι μήνες σε ένα χρόνο ή και σε δύο χρόνια είναι εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να έχουμε κάποια στοιχεία σε αυτήν την νομοθεσία, σε αυτές τις δύο δίδυμες, όπως είπα, οδηγίες, ε, κάτι το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μας με τον κύριο Άρημο και καταφέραμε νομίζω να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε για τους ε, καταναλωτές. Κάτι το οποίο δεν ήταν αυτονόητο ε, ευθύς εξ αρχής, γιατί επί τρία χρόνια έπρεπε να παλέψουμε για να περάσουν αυτά τα δικαιώματα. Και η Κομισιόν επίσης δεν συμφωνούσε πάντα. Και η δεξιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγκάστηκε να καταπιεί κάποια πράγματα, αλλά τελικά καταφέραμε να τα περάσουμε. Και με την βοήθεια ακούραστων συνεργατών κατάφερα να επιτύχω τον στόχο, τον οποίον είχα έναν στόχο ναι, για τον οποίο ε, πραγματικά με κορόιδευαν. Θυμάμαι ότι όταν είπα θέλω να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένα δικαίωμα σε κάποιο κράτος μέλος το οποίο θα μειωθεί λόγω αυτής της νομοσία. και μου λένε μα δεν γίνεται αυτή, δηλαδή θα κάνουμε πλήρη εναρμόνιση σε όλα τα, κράτη, τα κράτη-μέλη, δεν γίνονται αυτά πράγματα και όμω τα καταφέραμε. Καταφέραμε και σε συνεργασία με την ε, Επίτροπο να έχουμε αυτήν την ελάχιστη εναρμόνιση έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν οι φτάμενες διατάξεις και να ισχύουν. Γιατί οι λαϊκιστές βεβαίως θα χαιρόταν ε, αν κάναμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το οποίο πετύχαμε και νομίζω ότι είναι μια νομοθεσία προστασία των καταναλωτών άνευ προηγουμένου, η οποία προστατεύει ε, πάρα πολύ του καταναλωτέ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριο Άξελ Φω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε, κύρια Γκέπχαρτ, αγαπητή συνεισηγήτρια. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Κομισιόν για την πάρα πολύ προχωρημένη της ε, πρόταση που έγινε σε ένα νέο τομέα και να ευχαριστήσω και την κυρία Γκέπχαρτ για την εντατική αυτή συνεργασία που νομίζω οδήγησε τελικά σε κάτι καλό. Η κυρία Γκέπχαρτ ε, τόνισε την πτυχή της προστασίας των καταναλωτών. Εγώ ως ε, πιο δεξιός ε, ενδιαφερόμουν περισσότερο για το δίκαιο των συμβάσεων. Τελικά καταφέραμε να τα συμβιβάσουμε όλα αυτά και νομίζω ότι έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα. Ε, χρειάστηκε πολύ χρόνος βεβαίω, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα αφενός το τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων, με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και την μεγάλη αυτή συζήτηση που είχαμε για το τι θα γίνει με τα έξυπνα αγαθά, τα λεγόμενα, τα οποία καταφέραμε τελικά να περιλάβουμε σε αυτήν την ε, οδηγία και μετά στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με την έκθεση αριμών για τα απτά αγαθά θα έχουμε μια λογική ρύθμιση. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλαμε να επιτύχουμε ήταν μια όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη πλήρης εναρμόνιση σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και να μην αφήσουμε κενά παραθυράκια όσον αφορά τα έξυπνα αυτά αγαθά. Κάτι το οποίο βεβαίως οδήγησε στο ότι είπαμε ότι θα πρέπει οι συνέπειες και από τα δύο νομοθετήματα να είναι οι ίδιες, ανεξαρτήτως δηλαδή του εάν το ίδιο αγαθό το αγοράζουμε απευθείας, το παραγγέλνουμε στο διαδίκτυο ή το κατεβάζουμε. Και ε, συχνά εκεί πέρα ήταν οι δυσκολίες ε, και δυσκολευτήκαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Θεωρώ λοιπόν ότι τελικά δημιουργήσαμε μια καλή βάση για μια κοινή ψηφιακή εσωτερική αγορά από την ελάχιστη εναρμόνιση μέχρι την πλήρη εναρμόνιση στις ε, προθεσμίες παραδείγματος χάρη και Βεβαίω. Εντάξει, από το Συμβούλιο κάποιες φορές θα περίμενα κάποια πιο θετική αντιμετώπιση για το μέλλον, να θέλουν δηλαδή να δημιουργηθεί μια ψηφιακή εσωτερική αγορά και να μην επιμένουν ότι ο καθένας εδώ πέρα θα πρέπει να περιλάβει τον δικό του αστικό κώδικα και να λέει «Α, όχι, αυτό το πράγμα δεν αλλάζει». Όχι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επίπεδο στον ψηφιακό κλάδο όπου θα υπάρχει μια πανευρωπαϊκή εναρμόνιση γιατί αυτό είναι το σωστό. Η οδηγία την οποία εξετάζουμε σήμερα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάθεση των ψηφιακών περιεχομένων θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη ε, στιγμή λοιπόν έχουμε τις ελάχιστες απαιτήσει ε, με την οδηγία του 1999 και βεβαίως αυτό σημαίνει μία νομική ανασφάλεια η οποία υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτό το βήμα και θέλουμε να μην γίνεται πλέον καμία διάκριση το εάν δηλαδή οι υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά ή στο χύψη κράτος μέλος και υπάρχει αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως και έτσι σε κάθε κράτος μέλος πλέον είναι σαφής η νομική κατάσταση. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και θα προχωρήσουμε στο ψηφιακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους δύο συνεισηγητές. Πρώτης έκθεση, τώρα ο κύριος Πασκάλα Ρημό για τη δεύτερη έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, θα δανειστώ την παρομοίωση της κυρίας ε, Γκέπχαρντ, η οποία είπε ότι καταφέραμε μετά από μεγάλο αγώνα να γεννήσουμε δίδυμα. Εντάξει, εγώ δεν γέννησα βεβαίω, αλλά πραγματικά αισθάνομαι κι εγώ ως γονιό που έφερε κάτι στον κόσμο. Και βέβαια τα δίδυμα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά του πρώτους μήνες. Και αυτό ακριβώς καταφέραμε. Έχουμε αυτές τις δίδυμες οδηγίες, οποίες φέραμε στη ζωή. Και με αυτές τις δύο οδηγίες ε, έχουμε για πρώτη φορά ενιαίε εγγυήσει που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αγοράζει κανεί στο διαδίκτυο, είτε στον πραγματικό κόσμο, είτε μιλάμε για κάποιο υλικό αγαθό, είτε για μια εφαρμογή, είτε για ένα έξυπνο κινητό. Το έξυπνο κινητό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώ δεν ε, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μεταξύ κλασικών αγαθών και ψηφιακών αγαθών, γιατί πρόκειται εμπρότης για μια συσκευή την οποία μπορούμε να πιάσουμε με το χέρι, αλλά ταυτόχρονα περιέχει ένα λογισμικό και βεβαίως μπορούμε να κατεβάσουμε εκεί πέρα τις οποιασδήποτε εφαρμογές. Οπότε θέλαμε να έχουμε ενιαίες ε, διατάξεις ε, για την εγγύηση που θα ισχύουν και για τα παραδοσιακά θα λέγαμε αγαθά, αλλά και για μια εφαρμογή η οποία μας επιτρέπει να ακούσουμε ε, μουσική στο διαδίκτυο. Οπότε δεν θα θέλαμε ακριβώς να σταματήσουμε αυτές τις εφαρμογέ που κάνουν παραδείγματο χάρη video streaming. Επί της αρχής λοιπόν ισχύει το βασικό ότι ήδη με την αγορά υπάρχει ένα κλασικό αγαθό και ισχύουν κάποια πράγματα και για το ψηφιακό περιεχόμενο και για τις έξυπνες συσκευέ. Πρώτον, δηλαδή ότι όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση για αγαθά και περιεχόμενο. Δεύτερον, αν χαλάσει κάτι, μπορεί ο καθένας να ζητήσει επισκευή ή βελτίωση ή αντικατάσταση ή και λύση του συμβολέου. Όσον αφορά δε τα αγαθά, υπάρχουν κάποιες ε, πρωτοτυπίες εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την αντιστροφή του βάρους αποδοξιούς και τον διπλασιασμό της προθεσμίας αυτής, δηλαδή από έξι μήνες πάει στο ένα έτος και στα κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί αυτή η προθεσμία και στα δύο έτη. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα μετά από μία αντικατάσταση ή ε, επισκευή έχει την δυνατότητα ο καταναλωτής να λήξει την σύμβαση και να λάβει πίσω τα λεφτά του. Και τρίτον, αν διατηρεί την συσκευή για ένα συγκεκριμένο χρόνο ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να απευθύνεται στον κατασκευαστή για επισκευή ή αντικατάσταση. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα δικαιώματα τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτήν την ε, απλοποίηση και ενοποίηση θα κερδίσουν και οι επιχειρήσεις και μάλιστα οι μικρές επιχειρήσεις στο μέλλον δεν χρειάζονται να ασχολούνται με το ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν ε, όταν κάνουν μια εξαγωγή σε ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό ευνοεί κυρίως τους μικρούς ε, μπόρους που δεν έχουν νομικές υπηρεσίες όπως οι μεγάλες, τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα. Δίνουμε λοιπόν έτσι ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και δημιουργούμε ένα ενιαίο πλαίσιο στην εσωτερική ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν σε αυτό το κείμενο. Έδειξαν όλες οι ομάδες, όλες οι ομάδες την απαιτούμενη διάθεση για συμβασμούς και νομίζω ότι σε καιρούς πόλωση, όπου τα πάντα παρουσιάζονται ω άσπρο μαύρο είχαμε ένα χαρακτηριστικό θετικό παράδειγμα κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε εκ μέρου τώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το λόγο έχει η Επίτροπο Βέρα Γιώροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταπληκτική ευκαιρία που μας δίνετε, που μου δίνετε, γιατί μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα φτάνουμε τελικά στο τέλος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τις δύο αυτές προτάσεις που έχουν μια πολύ σημαντική προσθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους ε, ε, καταναλωτές και επιχειρηματίες. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε δύο δίδυμες εδώ πέρα προτάσεις. Η μία από τις προτάσεις αυτές ε, είναι πιο σύγχρονη η άλλη πρόταση ουσιαστικά έπρεπε να ακολουθήσει, αν θέλετε, τις όλες εξελίξεις για τις διαδικτυακές πωλήσει. Χρειάστηκε λοιπόν να ακολουθήσει την όλη διαδικασία της πρώτης πρότασης. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ θετική συνεργασία που είχαμε με τους συνομοθέτες και βέβαια να ευχαριστήσω τον, την κυρία Γκέπχαρα, τον κύριο Αριμόν και τον κύριο Φως, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζήσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές.